Okay, friends, we'll slowly start the meeting. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ε, όσοι από εσάς έχετε ξεχάσει την ε, κάρτα για τις ψηφοφορίες, μεριμνήστε παρακαλώ να την εξασφαλίσετε πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε. Σημείο 1 στην ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να την εγκρίνουμε χωρίς αλλαγές. Ωραία. Διερμηνία. Σε όλες τις γλώσσες πλην της Κροατικής. Διάλογος των εμπλεκομένων μερών. Εδώ αποφάσισαν οι συντονιστές να ζητήσουν η πρόταση για διαφανείς και με συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριληφθεί στον κατάλογο θεμάτων για τον διάλογο των εμπλεκομένων μερών για το 2016. Και έχει και η Γραμματεία επιφορτιστεί με την επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ υπό τον εισηγητή κύριο Καλβέ Σαμπό για να εντοπίσουν πιθανές ημερομηνίες και χώρο για το διάλογο. Στο 3 έχουμε μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα της συνεδρίασης της Επιτροπής. Δεν θα γίνει συνεδρίαση στις 16 και 17 Μαΐου Ανταυτού 14 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και Τρίτη 15 Μαΐου θα γίνει συνεδρίαση. Δευτέρα 3 με 6 και μισή. Τρίτη από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Εν εξελίξει δύο, οργανο συνομιλίες, εγκαθίδρυση ενός κοινού πλαισίου στατιστικών για τους ιδιώτες και τα νοικοκυριά επί τη βάση των δεδομένων σε ατομικό επίπεδο που συλλέγονται από δείγματα με τον κύριο Μέσεριτς εισηγητή. Ξεκινάει σήμερα ο τριμερής διάλογος και έτσι τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Έχετε τις κάρτες σας, τις έχετε βάλει στα μηχανήματα. Τροπολογία 13 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Επαληθεύουμε, 13. Πέρας. Απερίφθη. Με πέντε ψήφους διαφορά. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 προφορική τροπολογία, σοσιαλιστές και δημοκράτες, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 18 και 108 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 135 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη μάλλον. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αν ναι, έχει απορριφθεί, λέτε καλώς. Ελέγχουμε την 25. Άρχισε ψηφοφορία, πέρας και απεριφθεί όντως. Με τέσσερις ψήφους διαφορά. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές. Απερίφθη μάλλον, να επαληθεύσουμε την 30. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Με 6 ψήφους διαφορά εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 169 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 και 170 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη να επαληθεύσουμε τη 40 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας και απερίφθη με 7 ψήφους διαφορά συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παρακαλώ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μην συνομιλείτε. 45 υπέρ, κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε τις 45, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη με 6 ψήφους διαφορά, συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές. σας επαληθεύσουμε την 57. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη με ψήφους διαφορά. 4 και 58 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Κύριε Κώσα. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει αποσυρθεί η 58, αλλά φαίνεται ότι δεν ελευθεί υπόψη αυτό. Okay. We... Then we vote on Actually, we did, I didn't have that information. Όχι, δεν είχα την πληροφορία, κύριε Κώσα. Ψηφίζουμε την 4 πάντως, μόνο την 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε την 61 αρχής ψηφοφορία πέρας και απερίφθη με 14 ψήφους διαφορά τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ η 60 καταπίπτει. Πάμε στην 62. Απευθεία υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 66 υπέρ. Κατά. με συγχωρείτε λέει ο Πρόεδρος, 65 υπέρ, κατά, αποχές. Επαληθεύουμε την 65. Πέρα. Εγκρίνεται με 5 ψήφου διαφορά. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 67 απεριφθεί 68 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 7 και 75 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 86 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 σε δύο τμήματα έχουν ζητήσει οι σοσιαλιστές το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη λέω αλλά σε επαληθεύσουμε στην 11 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη με 10 ψήφους διαφορά. Δεύτερο τμήμα της 11 καταπίπτει. Και έτσι πάμε στην 85 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 και 92 μαζί ταυτόσιμες με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερο στην Επιτροπή της επασχόληση και των Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Και είναι 91 πίπτη. Και έτσι ψηφίζουμε την ε, πρόταση απόφαση του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε. Ή μάλλον όχι, θα την κάνουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Έχουμε δύο υπεραριθμούς από το ΕΛΚ. Εγκρίνεται 36 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, μία αποχή. Και πάμε στο σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος. 39 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχής εγκρίνεται. Ονομαστικά το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος στο σύνολό του. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται 34 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε τον εισηγητή. Άρα, τελειώσαμε το σημείο 4 και περνάμε στο σημείο 5, την έκθεση του κυρίου Κλόντο Χολάμ με θέμα την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας. Συμβαστική κάπα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική μια αλφα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νη. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 10 ψήφους διαφορά. Προχωράμε στη συμβαστική τροπολογία ε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία C. Τη βρήκατε. ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Είναι στη σελίδα 7 του καταλόγου ψηφοφορίας. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία β, β, περνάμε σελίδα 8, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία D. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και αυτή καταπίπτει. Και πάμε στην τροπολογία 40. Στη σελίδα 10 λέει πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία Ή μάλλον κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία J. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 62. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ ψηφίζει. Απορρίπτεται 31 ψήφι κατά. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63. 11. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία η 65 καταπίπτει. Πάμε στη 12. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Και 13 το ίδιο. Δεν, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 καταπίπτει. 73. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74 καταπίπτει. Τροπολογία 16 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και 75 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία L. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 82. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ κατά με ονομαστική κλίση για το σχέδιο έκθεση ψηφίζουμε για να είμαστε σίγουροι. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται με 41 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 7 αποχές. Τέλεια. Άρα, τώρα θα ψηφίσουμε την απόφαση να μπούμε σε ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις. είπε, κατά, αποχές. Α, ηλεκτρονικά πρέπει να γίνει. Ηλεκτρονικά στην κάνουμε τότε. Άρχεται η ψηφοφορία και τώρα λίγη. κρίνεται. 46 ψήφοι υπέρ. Άρα θα πάμε σε διαπραγματεύσεις διοργανικές. Και μέχρι τώρα πολύ καλή δουλειά έχει κάνει ο Κλοντ Γολά. Καταπληκτική σε ένα από τα θέματα που απασχολούν ε, και ε, την προεκλογική εκστρατεία ε, τις ευρωεκλογέ, όχι για ένα κόμμα μόνο, σχεδόν για όλα τα κόμματα. Αν θέλετε να ψηφίσει ο κόσμος στις εκλογές. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τους πολίτες. Πάμε λοιπόν στην ε, επόμενη έκθεση. Είναι το σημείο 6 στη μέση διαταξή. Έκθεση εφαρμογή στρατηγική Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής για την νεολαία του κυρίου Πιμέντα Λόπε. Συμβαστική 9. Ψηφί υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε και άλλη συμβιβαστική 6. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 63 κατά αποχές εγκρίνεται, τώρα 60, ορίστε. Θέλετε έλεγχο για την 63, παρακαλώ επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 30 ψήφι υπέρ. Προχωρούμε. Η τροπολογία 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές. Ας την ελέγξουμε αυτή παρακαλώ την 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με 28 ψήφους. 83 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ στην 101 ψηφίζουμε αρχίζει τώρα η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται με 29 ψήφους 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 105 υπέρ. Ορίστε. We check 104. The vote is... 104. Ηλεκτρονική παρήθευση αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται με 31 ψήφους. Ε, πάμε λοιπόν στην 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται τσεκ ωραία ελέγχουμε την 106 παρακαλώ αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και τελειώνει κιόλας Απορρίφτεται. με πέντε ψήφους διαφορά η τροπολογία τώρα 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 κατά τμήματα έχει ζητήσει η ομάδα των φιλελευθέρων, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Α, ας το λέξουμε παρακαλώ το δεύτερο τμήμα της 119 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και λίγη επίσης. Απορρίπτεται με 31 ψήφους κατά. Η τροπολογία 121 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά. Αποχές Ας την επαληθεύσουμε για καλό και για κακό. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Απεριφθεί. 28 ψήφια κάτω. Συμβιβαστική 1 τώρα. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 10. Ε, 9 ε, ναι, λέει η Πρόεδρος. Η τροπολογία ανακατέπεσε. Άρα, πάμε στην επόμενη σελίδα, στην τροπολογία 9. Ε, το ΕΛΚ έχει ζητήσει κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Ωραία. Θα ελέγξουμε το τμήμα υπαριθμό 2 της τροπολογίας ε, Ναι, αρχίζει τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Συνεχίζουμε. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 10. Ψήφι Κατά. Κατά. We δυστυχώς και πάλι χρειάζεται επαλήθευση. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 11 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές Θέλει έλεγχο η 12, παρακαλώ. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας τώρα. Εγκρίθηκε. Ε, ε, Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος. Στην 17 είμαστε, παρακαλώ, αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία και τελειώνει αυτή τη στιγμή. Εγκρίνεται 27, 21, 18 είπε, κατά αποχές. Την ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται με 28 ψήφους. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 29, αρκετά πιο κάτω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ, ωραία. Απολυφεύουμε την 33 παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και 2 εποχέ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον συντάκτη γνωμοδότηση. Προχωρούμε. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία, εξυγχρονισμός εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική FA ε, καταπίπτει αυτή. Οπότε θα προχωρήσουμε στη συμβιβαστική B, στην επόμενη σελίδα, ψήφιπε. Συμβαστικές, διορθώνει πρόεδρος, είπε κατά απόχες εγκρίνεται. S. Είναι στη δεύτερη σελίδα. Ξανά. Άντε. S, σίγμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική B, β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τσεκ. Ωραία, θα την ελέγξουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για τη συμβαστική B. Πέρασε. Εγκρίνεται με 28 ψήφους προς 20. Πάμε λοιπόν στην επόμενη τώρα συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική E ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. με τροπολογία 32 τώρα στη σελίδα 7 ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 44 ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική K υπέρ κατά Α, φόχες. Α, τσεκ. Συμβαστική και αρχής ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 25 ψήφους προς 22. Η συμβαστική 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Θέλετε έλεγχο χωρίστε. Στη 48 είμαστε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Απορρίπτεται 27-21. Προχωρούμε. Στη σελίδα 11. Ηλεκτροπολογία 61. Ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ φωνές. Ωραία, εγκρίν, ε, ε, ελέγχουμε συγγνώμη την 61. Αρχίζει τώρα η παληθεύση. Πέρας. Εγκρίνεται 27-20. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 75, σελίδα 13, το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 80, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική M, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Την επαληθεύουμε, τη συμβαστική M, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και τελειώνει. Με κρίνεται 28 ψήφι υπέρ. Προχωρούμε στην τροπολογία 91. Έχει και προφορική εδώ τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική Q υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική ο μικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 95 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απερίφθη το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο. Το δεύτερο τμήμα της 95. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is now closed. εγκριθηκε Εγκρίθηκε 28-19. Εγκρίθηκε με 28 ψήφους, τι θέλετε. Then we go to the third... Πάμε στο τρίτο τμήμα τώρα Τις 95 ψήφι υπέρ του τρίτου τμήματος. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. We go to amendment 100. Πάμε στην τροπολογία 100 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα πάμε στην τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική άρα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 133 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. «135 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται». Και τώρα είμαστε ήδη στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι αυτή και αρχιζει αμεσω αμέσως τώρα. Πέρας. Εγκρίθηκε 26-22. Ε, and thank you to the rapporteur, of course. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή φυσικά. Και τώρα, στο επόμενο θέμα, ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές. Αποσταθεροποιήθηκα ξαφνικά. ξαφνικά. Λοιπόν, ψηφίζουμε την συμβαστική 1, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. Συμβιβαστική 6. Αρχίζει η προφορία και εγκρίνεται με έξι ψήφους διαφορά. 31 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε. 31 Αρχίζει η ψηφοφορία.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 κατά αποχές απερίφθη 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 10 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε τη 10 αρχίζει πέρας 26 ψήφι υπέρ και εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 συμβαστική υπέρ κατά. Ας επαληθεύσουμε την 11. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται 27 ψηφοί υπέρ. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά και αρχίζει η ψηφοφορία και πέρας. Με 26 ψήφους εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. That means that we move to another very... Μπορούμε να περάσουμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα της σημερινής διάταξης. Το θέμα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Those of you who uh, won't stay to listen to the debate Παρακαλώ λίγη ησυχία για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση στα πλαίσια της έκθεσης για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και φροντιστές. Παρακαλώ, αν φύγετε από την αίθουσα, κάντε το αθόρυβα. Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα καλό κλίμα για τον εισηγητή, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Okay. Περνάμε αμέσω στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωής για τους γονείς και τους φροντιστέ. Θα δώσω το λόγο αμέσω στον εισηγητή μας, τον κύριο Κάζα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα σήμερα, τα Μαλτέζικα, μια και έχω την ευκαιρία. ασχολούμαστε εδώ και αρκετούς μήνες με την οδηγία αυτή και είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια ώστε να μεταφέρουμε αυτή την πολιτική από το ευρωπαϊκό στο περιφερειακό επίπεδο. Γιατί πρόκειται μια πολιτική που αγγίζει τους πολίτες και μπορούν να άμεσα να την κατανοήσουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υποβάλουμε αυτό το νομοθέτημα λίγο πριν τις ευρωεκλογές γιατί επηρεάζει τις οικογένειες των Ευρωπαίων. Στόχος της πρότασης είναι να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ της ε, ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής. Και ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το θέμα των ε, αδειών, γονικών αδειών, αδειών για παρέχοντες φροντίδα, κάτι που θα συμβάλλει στη βελτίωση και των εργασιακών συνθήκων τους και την εξισορρόπηση της ιδιωτική του ζωή με την επαγγελματική. Φυσικά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε σε θέματα απασχόληση και θα πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι πατέρε θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον δεκαήμερη άδεια πατρότητα, εγώ προτείνω να επεκταθεί αυτή η προθεσμία και σε περίπτωση υιοθεσία. και ανακαλύπτει όσου χαρακτηρίζονται πατέρε ή εξομοιώνονται με την ιδιότητα του πατέρα με βάση την εθνική νομοθεσία. Επίση, θεωρώ ότι η άδεια αυτή θα, είναι, θα πρέπει να είναι μεταποδοχών, όπω και η αναρωτική. Και θα πρέπει φυσικά να αντικατοπτρίζει την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει την άδεια το και θα πρέπει να δώσουμε ενάυσματα, να δώσουμε κίνητρα και στους πατέρες ε, για να αναλαμβάνουν ε, ισότιμα ε, τις ευθύνε της ανατροφής των παιδιών, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των επιπέδων αναρωτικών αδειών στα κράτη-μέλη, και της ευθυγράμμισης με την συγκεκριμένη άδεια. Επίσης, θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν μια αποζημίωση στο επίπεδο του 75% του ακαθάριστου μισθού και να μην είναι η βάση αναρωτική άδεια, για να μην υπάρχει ε, διαφορά μεταξύ των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την ηλικία, στο μέτρο που οι γονείς μπορούν να υποφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά, και μετά από ακροάσεις που είχαμε ενδιαφερομένους, και από τις δύο πλευρές, γιατί από τότε που ανέλαβα την έκθεση προσπαθώ να έχω εκτεταμένες διαβουλεύσεις. Μερικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η περίοδος της άδεια και άλλοι τη θεωρούν υπερβολικά φιλόδοξη. Δεν ήταν εύκολο να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των αντικρουόμενων απόψεων, αλλά είχαμε αρκετά καλή συνεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μερικοί ε, ενδιαφερόμενοι ανησυχούν και έτσι ε, εγώ μείωσα την επέκταση της ηλικίας από τα 12 στα 10. Σε ό,τι αφορά τους ε, παρέχοντας φροντίδα σε άλλα μέλη τη οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αποζημίωση, δικαίωμα αποζημίωση αντίστοιχα με πέντε ημέρες άδεια το χρόνο, με βάση την αναρωτική άδεια. Εγώ προτείνω μια τροποποίηση ώστε οι παρέχοντες φροντίδα να λαμβάνουν την ίδια αποζημίωση με τους ε, γονείς που λαμβάνουν άδεια γονική. 75% δηλαδή το καθάριστο μισθού ε, και αυτό να ισχύει για όλους άσχετα με, τη, με τις ρυθμίσεις της αναλωτικής στα κράτη-μέλη η οδηγία περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις που ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την δημιουργία κέντρων παροχής φροντίδας παιδιών ή να βελτιώσουν τις διατάξεις για τους παρέχοντες φροντίδα στην οικογένεια. Και εγώ προτείνω κάποια μέτρα για να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και χρειάζουν πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη και τη βοήθειά μας πολύ περισσότερο από τις μεγάλες ε, εταιρείε που έχουν περισσότερους πόρους. Γι' αυτό φρόντισα διατάξεις ε, της σχετικής νομοθεσίας να μην επιβαρύνουν επιπλέον είτε νομικά είτε οικονομικά τους, τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ ως συζητητής για την οδηγία αυτή θα φροντίσω να βρω μια σωστή ισορροπία και ένα αποτέλεσμα που θα εφαρμόζεται εύκολα και θα βοηθά, βοηθά όχι μόνο τους γονείς και φροντιστές αλλά και τους εργοδότες. Έτσι θα αφήσουμε ε, μια θετική εντύπωση και θετικό αντίκτυπο της οδηγίας για όλους, ώστε όλοι να υποφεληθούν από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εν κατακλείδη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησίγητες και τους συνεργάτες τους εννοείται, που ήταν πολύ υπομονετικοί μαζί μου και να ευχαριστήσω και τους δικούς μου συνεργάτες, γιατί είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι με τα μέτρα αυτά θα αφήσουμε πραγματικά το στίγμα μας και θα πειράσουμε σημαντικά την καθημερινότητα, αφήνοντας ένα πολύ θετικό αντίκτυπο από την, από την κοινοβουλευτική μας θητεία. Επίσης θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι το κοινοβούλιο είναι ισχυρό. Και καλό θα ήταν να να έχει νέα θέση στον τριμερή διάλογο για να μπορέσει να επηρεάσει την έκβαση και να έχει θετικές επιπτώσεις για όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Κύριε Κάσα, η Μαρία Αντριένα. Είναι σκιώδης, αλλά φαντάζομαι η κυρία θα λάβει τον λόγο. Εκ μέρους της παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μαρία Ρενά είναι όντως η σκιώδης αλλά ουσιάζει σε αποστολή αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν εκ μέρους της. Και ξεκινώ και εγώ, αλλά και εκ, και εκ όσο και προσωπικός με τις ευχαριστίες για την εξαιρετική δουλειά που έχει μέχρι τώρα κάνει για το θέμα αυτό. Να κοιτάξουμε τις τρεις βασικές αρχές της πρότασης. Την συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την καταπολέμηση της φτώχειας και ιδιαίτερος της δυσκολία ε, ε, στην επιβίωση για τις γυναίκες, αλλά και τα θέματα που έχουν να κάνουν με, τις παραδοσια... παραδοσιακούς ρόλους ε, για άντρες και γυναίκες. Με τις τρεις αυτές αρχές πιστεύουμε θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά επικοδομητικά μέσα σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων, διότι η προτάσεις ακριβώς αυτές τις ε, αρχές επιδιώκουν. Αρχές τις οποίες και εμείς ενστερνιζόμαστε. Καλωσορίζω τις τροπολογίες του εισηγητή για τη μη ε, μεταφερσιμότητα της ε, γονικής άδειας, τη δυνατότητα για εξασφάλιση εξωπρεπούς μισθού για τον εργαζόμενο όταν φεύγει σε άδεια ως γονέας ή ως φροντιστής. σε επίπεδο ε, αξιοπρεπές, όπως είπα, διότι η εξομοίωση, μείωση, εξίσωση αυτής της άδεια με την άδεια ασθενεία μπορεί να, είναι, να αποβαίνει βάρος του εργαζομένου. Είναι άλλωστε άνηση και η κάλυψη στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ορισμένα καλύπτεται με 60% ή 70% του ακαθάριστου μισθού, όπως το Γερμανία ή το Βέλγιο, ακόμα και με 20-30% του ακαθάριστου μισθού όπως στη Σλοβακία, ενώ σε άλλα κράτη μπορεί να καλύπτεται 100% μισθός. Και έτσι βεβαίως έχουμε και ένα αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορών συστημάτων. Επίσης, εάν διαφοροποιηθεί η γονική άδεια από την άδεια ασθενεία, θα έχουμε και ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο ότι θα αποκτήσει δική τη αξία αυτή η γονική άδεια. Δεν θα θεωρείται δηλαδή κάποιο είδου ασθένεια τον είναι κανεί γονέα. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική προσέγγιση στην κάλυψη αυτής της άδεια. Εδώ η πολιτική μας ομάδα λοιπόν πιστεύω ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει τις προτάσεις αυτές του εισηγητή. του άλλως και οι δικές μας προς το στόχο αυτών της κάλυψης της ε, γονικής άδειας. Τι Ο εισηγητής προτείνει ένα 70% με 75% επί του καθάριστου μισθού. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε κάπως πιο γενναιόδοροι και ως ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών και τι συμφωνούμε με την τεχνική προσέγγιση, δηλαδή την αντιμετώπιση των ε, ρυθμίσεων με διαφορετικό τρόπο. Είμαι βέβαια ότι μπορεί να διαφωνούμε ως προς τα ποσοστά τα ακριβή, αλλά θα βρούμε μια λύση. Δεν μπορούμε όμως να ακολουθήσουμε τον εισηγητή στο θέμα της αμοιβή της άδεια γέννησης. τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτή η γονική άδεια δηλαδή, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει πάντα να είναι μισθώσια η αποζημίωση. ειδικά για τους πατέρες. Εάν εξομοιωθεί με την άδεια ασθενεία που είναι στη Σλοβακία 20%, ποιος πατέρας από τη Σλοβακία θα ζητήσει άδεια για τη γέννηση του παιδιού του. Πρέπει να υπάρχει κάποια αξιοπρεπή κάλυψη. Και άρα θα πρέπει αυτή η άδεια γέννησης για τον πατέρα να ε, ευθυγραμμιστεί στην ε, γονική άδεια. Η Μαρία Ρένα πρόκειται να καταθέσει τουλάχιστον δύο τροπολογίες η μία σχετική με την ε, άδεια για τους πατέρες τη γέννηση των παιδιών τους, στον να Μια απλή αιτιολόγηση, δηλαδή να, εξε... εξασφαλιστεί η συμμετοχή του πατέρα στην ε, διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τρυφερή ηλικία και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί και η συμμετοχή τους στις δομές της οικογένειας για να ανατραπούν τα στερεότυπα Και επίσης ε, για το πεδίο εφαρμογής υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, γιατί η κυρία Ρενά θέλει να διευρυνθεί αυτό σε κάθε τύπο εργαζομένου και στους αυτοαπασχολουμένους και σε όσους εργάζονται σε ατυπικές μορφές εργασίας. Τρίτον, η κυρία Ρενά θέλει να υποστηρίξει την ε, ελάχιστη κάλυψη της μη υποβάθμισης λέει τη ρήτρα, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να υποβαθμιστούν οι ε, υπερεχόμενες από τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα προστασίες ε, καλύψεις. Και εδώ βεβαίως έχετε και το θέμα των ευέλικτων ε, διευθετήσεων στην εργασία και θα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων και οι ε, τα συμφέροντα των οικογενειών, δηλαδή μια εξισορρόπηση και των ενδιαφερόντων και συμφερόντων των εργαζομένων και των ε, διαφορών παραγόντων της οικονομικής ζωής. Ε, πάνω από όλα όμως πρέπει αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας να αποτελούν λύση επωφελή για τον εργαζόμενο, χωρίς να κινδυνεύει η οικονομική επιβίωση της οικογένειάς τους. Κοινό μα στόχο επίση είναι, ε, πιστεύω όλων, ε, να εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία σε επίπεδο κοινοβουλίου. Δεν είναι μόνο μια νομοθετική πρόταση αυτή η οδηγία. Δίνει ένα σαφέ μήνυμα για μια πιο κοινωνική και πιο η Ευρώπη, ύστερα από χρόνια λιτότητα που επευλήθησαν στους Ευρωπαίους πολίτες. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις λοιπόν στην Ευρώπη και σε αυτές συμπεριλαμβάνω και τον ξεβονίμων συνάδελφων θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Ριμπέιρο αντικαθιστά κάποιον, ζητεί το λόγο, όχι τίποτα από όλα αυτά. Α, η κυρία Μακεντάιρ, πίσω από την κυρία Ριμπέιρο. Α, δεν σας είδα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, γι' αυτό, μην νομίζετε ότι κρύβομαι πίσω από την κυρία Ριμπέιρο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η δικιά μας και οδησηγήτρια Γιάννα Σαντάσκα δυστυχώς απουσιάζει σήμερα και λυπάται γι' αυτό. Αλλά μου έστειλε την άποψή της να σας την πω εγώ και με μεγάλη μου χαρά να το κάνω. Λέει ότι αφού διάβασε προσεκτικά τις προτάσεις του εισηγητή χαίρεται που μπορεί να πει ότι έχουμε μια συναντήληψη για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, συμφωνεί με τον εισηγητή ε, της Επιτροπής Γυναικών, όπου τονίζει ε, τη σημασία να είμαστε ρεαλιστές και σόφρονες στα αιτήματά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίκαιρη πρόταση είναι και αξιόλογη και σημαντική. Ε, οι τροπολογίε τη ε, Γιάννα θα λάβουν υπόψη τα σε προβλήματα και ζητήματα. Πρώτον, να υπάρχουν υποδομές φροντίδας και φύλαξη των παιδιών. Πιστεύει η δική μα και ο συγκήτρια ότι είναι απολύτω κρίσιμο αυτό ε, για να ασκεί κανείς πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια και να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες στην αγορά εργασία. Βεβαίω, μόνο σε περίπτωση που θέλουν φυσικά οι γυναίκες και οι οικογένειες αυτές να το πράξουν. Επίσης, θα πρέπει να βεβαιωθούμε για τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτά στις επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό και πραγματικά ο εισηγητής το έχει λάβει υπόψη στις τροπολογίες του. Γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά είναι γεγονός ότι ε, ορισμένες ευέλικτες μορφές εργασίας μπορεί να επηρεάσουν πολύ μικρές εταιρείες με τρόπο έδικο Και η τελική μας ε, πρόταση θα πρέπει αυτό να το αντανακλά. Επίσης, η σκιώδη συγγήτρια μας ε, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές στις περιπτώσεις που οι γονείς έχουν παιδιά με αναπηρίες και προτείνει ο συγγητής όταν ζητούν ευέλικτες μορφές εργασίας να αρχίζει από χαμηλότερη ηλικία, μικρότερη ηλικία του παιδιού και η δικιά μας συζητήτρια το βλέπει αυτό θετικά ε, εν ώψη ενός μελλοντικού συμβιβασμού. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών για παιδιά με αναπηρίες και ε, ειδικές ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας για να θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ε, κατάσταση των φροντιστών τώρα και θα καταθέσει ε, τροπολογίες και προτάσεις ε, για να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες διευθετήσεις και θέσεις των άτυπων φροντιστών μελών της οικογένειας. Αυτά από την εισηγητριά μας. Να αναφερθώ τώρα και λίγο στη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου διότι διαφέρει. Θα είναι τελείως νέα μία αξίωση για άδεια φροντιστού. Υπάρχει όμως ε, πολλή νομοθεσία χώρια στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, που καλύπτει τις διατάξεις που προτείνει η οδηγία. Άδεια πατρότητας, ε, με απολαβές, γονική άδεια, ευέλικτες μορφές εργασίας κτλ. Οι δικέ μου λοιπόν ανησυχίες ποιες είναι ότι η πρόταση θα μπορούσε να προσκρούσει σε κείμενο δίκαιο, καλά ανεπτυγμένο και λειτουργών σε, αυτή τη σε αυτό το... το θέμα, σε αυτό το πεδίο. Δεν υπάρχει κατοχυρωμένο δικαίωμα για τους φροντιστές σήμερα που να το διεκδικούν. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ε, ε, ανάμεσα σε πολιτικές που υπάρχουν και λειτουργούν σωστά και εκείνες που θέλουμε να νομοθετήσουμε, έτσι ώστε να φτάνουμε στο πραγματικό μας στόχο. Θέλω όμως και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Βέμπερ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί ήταν πολύ σοφή και συνετή προσέγγιση του και κυρίω η επιδίωξή του για ευρεία σε πλειοψηφία η συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η ενότητα θα είναι σημαντική αν θέλουμε να έχουμε θετικό για μας αποτέλεσμα στον τριμερή διάλογο, γιατί γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων ε, και πολύ μεγάλη διαφορά από εμά και από αυτά που συζητούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σίγουρα τη συζήτηση της ισορροπίας ε, ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής είναι αδύνατο να μην σκεφτόμαστε και την αδιαμητρότητα. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το προσπαθήσουμε να την αφήσουμε κατά μέρο προς το παρόν. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σοφή προσέγγιση, πολύ συνετή, να μην την εξώσουμε με την αναρωτική άδεια, αλλά να ε, θεσπίσουμε ένα ενιαίο ποσοστό 70-75%. Εμείς συμφωνούμε με το 75%. Γνωρίζουμε ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι το 85% του ακαθάριστου μισθού είναι αυτό που προτιμούν γενικώ οι άνδρε προκειμένου να διεκδικήσουν την άδεια πατρότητα. αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προ διαπραγμάτευση το συγκεκριμένο ποσοστό, το ίδιο του ποσοστού. Με εκπλήσει ότι στις πολυάριθμε συναντήσεις που έχω, όπω και οι συνάδελφοι φαντάζομαι για το θέμα αυτό, πολλοί αντιμετωπίζουν την εγκυμοσύνη σαν κάτι που έχει πολύ σύντομη διάρκεια ενώ διαρκεί εννέα μήνες, πολύ λίγο λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, μας δίνει χρόνο να προετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται. Δεν γίνεται εν μία νύχτη. Ούτε ε, ε παρετείται κανείς ή βγαίνει σε άδεια εν μία νυχτή. Μπορεί να τα προβλέψει όλα αυτά. Και αυτό ισχύει και για τι μητέρε και για του πατέρε και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μπορεί να γίνει ένα καλό προγραμματισμό για να μην παρεμποδιστούν οι δραστηριότητε μια επιχείρηση. Γι' αυτό όμω θα πρέπει να γίνει συζήτηση, προεργασία, καλή διαπραγμάτευση και μπορούμε να βρούμε λύση. Σίγουρα με τι τροπολογίε μα θα ταχθούμε υπέρ τη ιδέα ελαστικών αριθμίσεων για την εργασία. Και νομίζω σε αυτή την ελαστικότητα θα ανθίσει το μέλλον της αγοράς εργασίας με καλύτερη συζήτηση και συνεννόηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης, ε, είμαι υπέρ και μάλλον θα καταθέσω και σχετική τροπολογία για τη συμπερίληψη και των αυτοαπασχολουμένων και όλων των ειδών ε, εργαζομένων, γιατί είναι λογικό να ισχύει και για αυτούς η άδεια. Επίσης, ε, θα ζητηθεί δεσμευτική εφαρμογή της άδειας πατρότητας. Εδώ έχω αρκετέ αφιβολίε για το αν μπορούμε να είμαστε τόσο φιλόδοξοι και τόσο υπερβολικοί. Μπορούμε έτσι να ε, καθορίσουμε κάποιες συμπεριφορές, να προσδιορίσουμε κάποιες συμπεριφορές ή να τις καλουπώσουμε, αλλά καλύτερα να το συζητήσουμε περαιτέρω στη διαπραγματευτική διαδικασία. Και ε, για την παράταση του ηλικιακού ορίου μέχρι τα 12 να ισχύει για, για παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Αυτό έχει νόημα. Ε, ή να μείνει στα 10, να μην έχουμε ούτως ή άλλως διεύρυνση. Αυτό θα το συζητήσουμε επίσης, θα το διαπραγματευτούμε και, και, το, και τη διάρκεια της διασπατρότητα. θα, θα πρέπει να τη διαπραγματευτούμε, γιατί στο Συμβούλιο είναι πολύ σκληροί και θέλουν περιορισμό της διάρκειας ε, όσο γίνεται. Πάντω εμεί είναι σημαντικό στην Επιτροπή Απασχόληση να έχουμε ισχυρή εντολή προ τον εισηγητή μα για τι περαιτέρω διαπραγματεύσει. Γιατί αν και εμεί είμαστε διχασμένοι θα είναι πολύ πιο δύσκολη και αποδυναμωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι περαιτέρω συζητήσει με το Συμβούλιο. Και α ευχηθούμε καλή τύχη. Η Τάινια Γκονσάλες Πένια, εκ μέρους τη Γκουέ και οδηγητρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον γιατί για τη δέσμευση, την αφοσίωσή του, την ε, εργασία του και τις εξηγήσει που μας έδωσε τώρα και την ε, εστίαση, τον προσανατολισμό του σχεδίου έκθεσης. Θέλω να σας αναφέρω τρία σημεία που τα βρίσκω σωστά. Πρώτον, ε, η αναφορά στις υποδομές φροντίδας. Έλειπε αυτό από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς θα προσπαθήσουμε από την ομάδα μας να κάνουμε τροπολογίες για να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Είναι εκ των Κάνευ για να επιτύχουμε την ισότητα στην αγορά εργασίας. Επίσης πρέπει και ο δημόσιος τομέας να απτυχθεί πολύ περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, χαιρόμαστε που ε, διατήρησε στο ακέραιο μη δυνατότητα μεταβίβασης της γονικής άδειας ακριβώς για να υπάρχει πιο ισότιμη ε, συμμετοχή και στην αγορά εργασίας αλλά και στην ευθύνη ε, της ανατροφής. Και το τελευταίο είναι το ποσοστό για το καθάριστο μισθό για την ε, φροντίδα να εξώνεται με την αναρωτική άδεια, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις διάφορες χώρες μέλη, ακριβώ για να έχουμε την εγγύηση ενός ε, αξιοπρεπούς ε, ποσοστού. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να έχει δείξει έκθεση μεγαλύτερη φιλοδοξία, πέντε τον αριθμό. Πρώτον, το συγκεκριμένο ποσοστό που αναφέρεται, 75% του ακαθάριστου μισθού για την αποζημίωση ε, των ε, ε, αδειών, των γονέων και των φροντιστών, το θεωρώ αυτό ανεπαρκές. Διότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αμοιβέ είναι σε ευθεία αναλογία ε, με την άδεια που παίρνουν οι πατέρες, δηλαδή αν ξεσωθεί πλήρως 100% ε, παίρνουν όλο τους το μισθό, ε, θα παίρνουν την άδεια αυτή περισσότεροι οι πατέρες και θα συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική κατά την άποψή μου η άδεια αυτή πατρότητας. Αναγνωρίζετε λοιπόν ότι είναι ισότιμοι άνδρες με γυναίκες και ε, δύο εβδομάδες ε, για το τοκετό, για την υιοθεσία ε, και τα λοιπά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Τρίτον, δεν βλέπω τροπολογίες για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουν διαγραφεί κάποιες αναφορές από το κείμενο σχετικά. Εμείς θεωρούμε ότι ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να απορρίπτει τα αιτήματα των εργαζομένων. Δεν είναι στη διακριτική τους ευκαιρία, είναι δικαίωμα. Και το δικαίωμα αυτό μπορεί να το διεκδικήσει και να κάνει χρήση του εργαζόμενου να το επιθυμεί η εργαζόμενη. Δεν είναι στο χέρι τη επιχείρηση να το αποφασίζει, να το απορρίπτει. Επίση, ε, έγιναν και πολλέ αναφορέ και υπενιγμοί για τι μικρομεσαίε, μεσαίε, μικρέ, πολύ μικρέ επιχειρήσει. Ε, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά και όλοι μπορεί να ανησυχούμε, αλλά στη μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάνηκε ότι υπάρχουν ε, ωφέλειες για την απασχόληση και την ανάπτυξη μέσω μακροπρόθεσμα. Και μπορεί στην περίπτωση των γυναικών ε, εγκαίρως οι επιχειρήσεις να οργανώνονται για να δίνουν τις άδειε, ενώ για τους ε, άντρες δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο που θα έπρεπε. Και ε, τέλος, δεν κάνετε λόγο για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις ιδιαιτερότητες σε περίπτωση ε, πολλαπλών γεννήσεων και για τους φροντιστές δεν αναφέρεστε σε μέλη της οικογένειας δευτέρου βαθμού. Κατά την άποψή μου και το έχω πει πολλές φορές, είναι λάθος η εστίαση που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη σε αυτή την έκθεση, ε, στην οδηγία για τη μητρότητα. Δεν είναι μόνο η μητρότητα, είναι και η πατρότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο και από κοινού. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και αυτά. Ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βελτιώσουμε και πιο ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μητροφάνος, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Κάσα για τη δουλειά του, την προσπάθεια για βελτίωση του εγγράφου που μας ε, υπέβαλε η Επιτροπή. Η Ντανούτα, η ε, ε, συνάδελφος και πρώην μέλος της Επιτροπής μας, Έχει ήδη κάνει πολλή δουλειά για το έγγραφο αυτό, ώστε να μετατραπεί σε ένα καλό κείμενο ε, για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Έχει ξεκινήσει το 2016, εγώ θα συνεχίσω αυτό το, αυτή την προσπάθεια στην ίδια γραμμή. Συμφωνώ με, την, με τον εισηγητή ότι ίσως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βέβαια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Ωστόσο, θα ήθελα να δώσω μια διαφορετική προοπτική, γιατί η προτεραιότητα είναι ο εργαζόμενος και η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Δεν ξέρω πόσο επιλύονται με τις προτάσεις ε, τα προβλήματα του συνδυασμού αυτής της ισορροπίας στο έγγραφο. Ιδιαίτερη δε προσοχή θέλω να δοθεί στο επίπεδο της αποζημίωσης για αυτήν την άδεια. Γιατί στο αρχικό κείμενο λέγεται ότι το επίπεδο των επιδομάτων θα πρέπει να είναι ισοδύναμο τουλάχιστον μετά όσα θα εισέπρατε σε περίπτωση άδεια ασθενεία ο εργαζόμενος. Αλλά η κάλυψη στο επίπεδο της ε, άδεια ασθενεία για μας δεν είναι ικανοποιητική είναι διαφορετική σε πολλά κράτη-μέλη η αποζημίωση άδειας ασθενείας μέχρι και 40% μπορεί να φτάσει, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επιδόματα σε αυτό το επίπεδο. Εμείς θα θέλαμε να καλυπτούνται πλήρως τα επιδόματα και οι ελάχιστε προδιαγραφέ για την πατρική άδεια μπορεί να εμφανίζονται στην πρόταση της Επιτροπής, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, θα θέλαμε να υπάρχει πλήρης κάλυψη με το μισθό. Η πρόταση της Επιτροπής για την αύξηση της ηλικία για την, του παιδιού μέχρι τα 20 χρόνια μας βρίσκει σύμφωνος και δεν συμφωνούμε με τη μείωση της στα 10 χρόνια, όπως προτείνει ο Είχαμε ήδη κάποιες επαφές με ενώσεις εργαζομένων, εργοδοτών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες ως προς το ζήτημα της ηλικία των παιδιών, αλλά για μας μόνο θετικά μπορεί να φέρει, γιατί το να μιλάμε μόνο για την μικρή παιδική ηλικία. μπορεί να οδηγήσει προβλήματα στην παραγωγικότητα. Ενώ αν εξαπλωθεί σε όλη την ε, ηλικία του ανήλικου μέχρι και τα 20 χρόνια αυτή η άδεια, θα μπορέσει να εξισορροπήσει καλύτερα την παραγωγικότητα και θα φέρει μόνο πλεονεκτήματα. Θα καταθούν σχετικές τροπολογίες. Επίσης, το αρχικό κείμενο της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη επαρκώς τις ε, ανάγκες των φροντιστών. Θα πρέπει να υπάρχει των ε, γονέων που μόλις ανατρέφουν ε, τέκνα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια σχετική ρύθμιση. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι ήδη υπάρχει σχετική νήξη στο κείμενο της Επιτροπής για την περίοδο δε των πέντε ημερών ε, για τον φροντιστή δεν θεωρούμε ότι είναι αυτό μια άδεια για φροντιστή και θα θέλαμε να αυξηθεί η σχετική περίοδος. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Η Λάουρα Οτζή από το EFTT ε, δεν είναι παρούσα. Μήπως την αντικαθιστά κάποιος. Ούτε η Ζωέλα Μελά αντικαθίσταται. Όχι. Οπότε περνάμε στους λοιπούς ομιλητές. Ο κύριος Κώσα πρώτος. Ευχαριστώ πολύ ε, που μου δίνετε το λόγο. Ε, κυρία Πρόεδρε, έχω πολλά να σας πω. Να μοιραστώ μαζί σας ε, πολλές σκέψεις. Το σχέδιο της έκθεσης είναι ένα εξαιρετικό κείμενο καταρχάς και ε, πραγματικά είναι πολύ καλή βάση και κίνητρο για κοινό προβληματισμό. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Ε, εξαιρετική δουλειά έχει κάνει ο εισηγητής για να συνδυάζει κανείς καλύτερα την επαγγελματική με την ιδιωτική ζωή. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολείται με την οικογενειακή πολιτική. Αυτό όμως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την αρχή της επικορικότητας και την αρχή της αναλογικότητας εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως σας είπα και προηγουμένως και σε άλλες ευκαιρίες, έχω κι εγώ επιφυλάξεις ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που ακούσαμε προηγουμένως από κάποιους συναδέλφους. Στη μελέτη αντικτύπου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εξετάζεται επαρκώς ο αντίκτυπος σε πολύ μικρές εταιρείες που έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και χαίρομαι που ο εισηγητής επικεντρώνεται πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Επίσης πιστεύω ε, ότι έχει μεγάλη σημασία το σύστημα να γίνει πιο ευέλικτο δεν επιθυμούμε να αναγκάσουμε κανέναν να επιλέξει μεταξύ επαγγέλματος και οικογένειας. Ευελιξία μπορεί να υπάρξει, για να δούμε ποιες λύσεις προτείνονται. Και θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κρίμα να μειωθούν, να περιοριστούν οι οικογένειες στην Ευρώπη εξ αυτού του λόγου θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές εμπειρίες με τις άδειε τις γονικές. Έχουν εμπειρίες τα κράτη-μέλη και υπάρχουν και χώρες που δίνουν πολλά χρήματα ε, και αμείβουν τη γονική άδεια και για τους πατέρες, αλλά λίγοι πατέρες επιλέγουν να ε, αξιοποιήσουν αυτό το χρονικό διάστημα. Στην Εσθονία είναι η αποζημίωση 100% του μισθού. Και μάλιστα μπορούν να παραμένουν 18 μήνες στο σπίτι οι πατέρες για να φροντίζουν τα παιδιά τους. Ε, σε άλλα κράτη-μέλη είναι αποζημίωση το 10% του μισθού. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί τέτοιες μεγάλες διαφορές από 10% σε 100% είναι τεράστια η ψαλίδα. Θα πρέπει από κοινού να το κοιτάξουμε, να δούμε ποιος κάνει λάθος. Και πώς μπορούμε να δώσουμε νέα κίνητρα και να παροτρύνουμε. Ε, τους ε, πατέρες. Να πω δύο λόγια τώρα για την οικογενειακή πολιτική που ε, ακολουθεί η Ουγγαρία. Είναι καλό το γεγονός ότι μπορούν να μένουν πολύ καιρό στο σπίτι οι γονείς για να φροντίζουν τα παιδιά τους, αλλά δεν πρέπει να έχουμε μεγάλες απώλειες εισοδήματος. Λοιπόν, ε, δεν το λέω αυτό επειδή είμαι Ούγγρος, αλλά κοιτάξτε λίγο και τι κάνει η Ουγγαρία. Ε, ε, μ' αρέσει πολύ το, το εσθονικό σύστημα, 18 μήνες με 100% του μισθού για τους πατέρες για να ε, μπορεί να ανατρέφει και ο πατέρας το παιδί του. Και υπάρχουν και πολύ μεγάλα επιδόματα τέκνων. Δεν λέω να είναι 18 μήνες απολύτως, αλλά έστω και 6 μήνες να είναι, αλλά να μπορούν ε, οι γονείς να επιστρέφουν κιόλας κάποια στιγμή ε, στο χώρο εργασίας τους. Οικονομική υποστήριξη λοιπόν δεν είναι το παν. Θα πρέπει να βελτιωθούν και υποδομές ε, φροντίδας και φύλαξης των παιδιών, δηλαδή να υπάρξει και ένα σύστημα ολόκληρο που να υποστηρίζει τους γονείς. Και καλό θα ήταν να το κοιτάξει και αυτό ο εισηγητής. Ε, θα είχα και θα κάνω τροπολογίες, γιατί αν επεκταθεί αυτό το σύστημα και το σύστημα φύλαξη των παιδιών, αυτό είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για την οικογένεια. Και χάρηκα για τα σχόλια που άκουσα για ε, την υποστήριξη των γονέων ε, με παιδιά με αναπηρίες στην Ουγγαρία οι γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες έχουν περισσότερη άδεια. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερη φροντίδα. Άρα έχουν και περισσότερα βάσανα αυτές οι οικογένειες. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του και χαίρομαι ε, για τις μελλοντικές συζητήσεις και συνεργασία που θα έχουν. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ριμπέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Νταβίτ Κάσα για το έργο του. Γιατί ήδη έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχει ακόμη μεγάλη δουλειά μπροστά του για να βρει την επιθυμητή ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών απόψεων. Γιατί είναι σημαντικό, παρά τις κριτικές, να έχουμε αυτή την επιτυχία στην ε, κοινοβουλευτική μας θητεία, γιατί όλα τα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών είναι στραμμένα πάνω μας. Ε, δεν πρέπει να επεκδηθούμε των ευθυνών μας. Είμαστε οι ε, νόμοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, εμείς οι Ευρωβουλευτές. Θα πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε το δικό μας έργο μας θέση από τη θέση του Συμβουλίου. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι οικογενειακές ευθύνες δεν εξαντλώνται με την γέννηση των παιδιών. Το θέμα της ε, ε, πατρότητας είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει και οι πατέρες να αναλαμβάνουν με των ευθυνών. Θα πρέπει και οι δύο γονείς ε, να μοιράζονται τις ευθύνες, αλλά όχι μόνο στην πρώτη φάση της γέννησης, σε όλες τις φάσεις της ζωής που χρήζει κάποιες φροντίδας. Ε, τα παιδιά αρρωσταίνουν, φυσικά δεν είναι όλες οι είδες, αλλά χρειάζεται μία φροντίδα το παιδί που έχει γρήπη, αλλά πολύ διαφορετική φροντίδα χρειάζεται ένα παιδί που θα πρέπει να ε, νοσηλευθεί γιατί έχει καρκίνο ή μία σοβαρή ασθένεια. Επίσης, έχουμε παιδιά με αναπηρία έχουμε ηλικιωμένους ε, γονείς που θα χρειαστούν επίσης φροντίδα. Ε, και μάλιστα αυτό το φαινόμενο θα επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο που γυράσκει ο ευρωπαϊκός πληθυσμό. Γι' αυτό χρειάζεται η οικογενειακή υποστήριξη για τα πιο ηλικιωμένα μέλη τη οικογένεια. Οπότε σε αυτό το έγγραφο θα πρέπει να υποβάλουμε μια πρόταση που δεν θα εξαντλείται στο ζήτημα της ε, άδεια της γονικής ή της άδεια πατρότητας, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που θα επιτρέψουν την εξορρόπηση μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού ιδιωτικού βίου, χωρίς διάκριση μεταξύ των δύο φύλων, χωρίς ε, να επιβαρύνεται με τη φροντίδα των μελών ε, της οικογένειας των Χρυσό Βοήθεια μόνο η γυναίκα και φυσικά να έχουμε μια ενιαία ε, ρύθμιση για την αμοιβή των αδειών αυτών και για το επίπεδο τους. Ο κύριος Γκέρικε. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον Ντοβιτ Κάζα. Το γεγονός και μόνο που ακούμπησε το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Το πρόβλημα όμω είναι ότι δεν έχει, καμία, δεν έχει βρει τη θέση της ε, στην έκθεση αυτή η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής ιδιωτική ζωή για τους ε, γονεί. Τι είναι αυτό δηλαδή που μας λέτε, ότι περιγράφεται ως, χώρος, ως χρόνος διακοπών η γονική άδεια. Αυτό είναι ντροπή, είναι προσβολή γιατί η μητέρα, το πατέρα ή οποιονδήποτε άλλον φροντίζει κάποιον. Τώρα είναι κανείς γονιός. Σημαίνει με πολύ διαφορετικούς τρόπους ότι μπορεί να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του αν το παιδί του είναι άρρωστο. Σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση πάντα να δουλεύει σε πλήρη απασχόληση, αναγκάζεται να προσφέρει μερική μόνο εργασία. Σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής του έχει και έλλειμμα στη σύνταξη. Γιατί, Γιατί δεν αναγνωρίζεται ως εργασία η υπηρεσία που προσφέρει ο γονιός. Εάν αυτό δεν γίνει, δηλαδή αν δεν αναγνωριστεί ως χώρος χρόνος εργασίας, η φροντίδα για τα παιδιά, όπως συμβαίνει για το βρεφονιπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και το καθεξής, τότε θα παραμείνει το κενό. Και η ισορροπία δεν πρόκειται να εξασφαλιστεί με τίποτα. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να ταξινομηθεί η περίοδος της φροντίδας για τα παιδιά και πώς. Για σκεφτείτε να μπορούσαμε στα 27 κράτη-μέλη να παίρναμε μία ε, ε, εικόνα του τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν οι βρεφονιπιακοί και η παιδική σταθμοί για να ε, αντλήσουμε από εκεί ένα γνώμονα για το πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση για το γονιό που φροντίζει το παιδί του. Και μετά και σε όρους απασχόλησης και ε, μισθολογικούς το πιο αλλά και φορολογικού όρου, το πιο συμφέρον είναι να μην κάνει κανεί παιδιά. Σε όρου φορολογικού, σε όρου μισθολογικού, σε όρου απασχόληση είναι και σταδιοδρομία είναι καλύτερο να μην κάνει κανεί παιδιά. Λοιπόν, όσο ισχύουν αυτά, δεν πρόκειται να μπορούμε να κάνουμε λόγο για ισορροπία μεταξύ οικογενειακή ζωή και επαγγελματική. Σε δημοσιονομικού όρου, λοιπόν χρειάζεται να ε, δοθεί μια εύνοια κίνητρο για όσου έχουν παιδιά. Και αν κοιτάξουμε τι σημαίνουν ανάγκες των παιδιών, αν θέλουμε να ε, προσανατολιστούμε στις ανάγκες των παιδιών, αν διανοηθούμε τι χάνουν τα παιδιά εάν δεν μπορεί ο γονιός τους να τα φροντίσει, τι είδους, ε, και μάλιστα ανάλογα με την φάση της ηλικίας την οποία παίρνουν. Τα δύο πρώτα χρόνια πρέπει ο γονιός να είναι συνέχεια παρόν. Ε, αυτή είναι η πρώτη φάση, από τα, από τα 3 έως 6 χρόνια, μετά έχουμε μια δεύτερη φάση από τα 7 έως τα 12 χρόνια, για, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι, ανάλογα με την εξέλιξη του παιδιού. Και εδώ πάλι θα πρέπει να γίνει σχετική προσαρμογή του συστήματος για να καλυφθεί και οικονομικά η ε, παροχή της υπηρεσίας του γονιού. Μόνο όταν μπορούμε να το κάνουμε αυτό θα μπορούμε να μιλούμε για ισοδίκαιη αντιμετώπιση ώστε να μην αντιμετωπίζουν οι γονείς. Και εδώ δεν διακρινώ μεταξύ μητέρα ή πατέρα ε, έλλειμμα ως προς τη σύνταξή τους στην, ε, στο τέλος της αδειοδρομία τους και της ηλικία τους. Ε, φυσικά θεωρώ ότι η μητέρα πρέπει να είναι παρούσα συνεχώς τους έξι πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού, αλλά μετά μπορεί ο πατέρας οπωσδήποτε να αναλάβει και 100% ακόμη την μέρημνα για το παιδί του. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι θετικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή μας με την έκθεση του κυρίου Κάζα θα εμπλουτίσει το, την πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και επίσης είναι και πολύ δύσκολο και μακροπρόθεσμα ε, δημιουργείται ένα δίλημα γιατί προσπαθούμε να συνδέσουμε πράγματα που είναι ασύνδετα μεταξύ τους και όμως φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να το επιχειρήσουμε. Γιατί θα, καλό θα είναι να μπορεί κανείς να έχει επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομή και ταυτόχρονα να είναι ευτυχισμένο στην ιδιωτική του ζωή. Είναι κάτι τέτοιο ρεαλιστικό μπορούμε να το επιτύχουμε. Και μόνο η έννοια της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματική και της ιδιωτικής ζωής σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια ισότιμη κατανομή μεταξύ του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου. Ενώ υπάρχει συνήθως μια δυναμική ισορροπία στον κόσμο, δεν είναι 50-50, ε, δεν υπάρχει απόλυτη ισορροπία, υπάρχει μια δυναμική. Και παντού ισχύει αυτό. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε η οικογένεια ή ο επαγγελματικός βίος έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες. Και παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην Ευρώπη 65% των πτυχιούχων ανωτέρων ε, ιδρυμάτων είναι γυναίκες, αλλά απασχολούνται κατά 12% λιγότερο από τους άνδρες, οπότε υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μεν αποφυτούν και έχουν πτυχία, αλλά δεν δουλεύουν τόσο πολύ όσο οι άνδρες. Οπότε καλό το έγγραφο και θα πρέπει να το εμπλουτίσουμε όσο μπορούμε, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουμε α, αν είναι απαραίτητο μια ευρωπαϊκή οδηγία να αποκαταστήσει την ευτυχία ή την, να συνδυάσει την ευτυχία στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή. Κανονικά Κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να μεριμνά για να εφαρμόζει συγκεκριμένες αξίες και αρχές που θα επιτρέπουν ε, ισότητα των φύλων ε, σε τέτοια σημαντικά θέματα. Η πρόσβαση στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, σε κέντρα αφροντίδας, στήριξη από τους εργοδότες, με προγράμματα ενίσχυσης της εταιρείας σε περίπτωση που φεύγουν σε άδεια πατρότητας ε, οι υπάλληλοι. Επίσης, ε, τι γίνεται με παιδιά με αναπηρίες ή με γονεί που πρέπει να φροντίζουν ηλικιωμένου ε, γονεί, ηλικιωμένα μέλη τη οικογένεια που χρήζουν φροντίδας. δεν είναι τα ίδια τα είδη φροντίδας μεταξύ παιδιών και ηλικιωμένων. Θα πρέπει να υποχρεώνουμε τον πατέρα να βγει σε άδεια ενώ είναι πολύ σημαντικό να μένει η γυναίκα και να θυλάζει τους πρώτους μήνες και παρόλα αυτά να υποχρεώσουμε τον πατέρα να βγει σε άδεια πατρότητας. Και στην Πολωνία έχουμε ε, το πρόγραμμα 500 συν, ε, που, ένα επιπλέον επίδομα που προβλέφθηκε για τα παιδιά. Επίσης, ε, ένα οικογενειακό επίδομα που δίνεται από το κράτος για τους βερφονιπιακούς σταθμούς και θα θέλαμε να γίνεται και δωρεάν κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα για τα παιδιά με αναπηρίες. Επίσης, έχουμε επιδόματα για στεγαστικά ώστε να εξασφαλίσουμε στέγαση και πρόσβαση στην ε, κατοικία και σε νέους. Πρόκειται για δράσεις που αυτόματα διευκολύνουν το συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Φοβάμαι ότι ε, καλό είναι να το κάνουν τα κράτη-μέλη ε, ξεχωριστά και πιστεύω ότι είναι δύσκολο να το κάνουμε με το στανιό, με μια ευρωπαϊκή οδηγία. Θα πρέπει τέτοιες επιχειρηματολογίες ε, δεν ευσταθούν. Ναι, είμαστε υπέρ της εξισορρόπησης, αλλά καλύτερα σε εθνικό επίπεδο τα μέτρα. Ο κύριος Πιμέντα Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το έργο του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία που στόχο έχει την συμφωνία και την έγκριση της οδηγίας αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε κάτι που γνωρίζουμε ήδη για την ε, θέση και τις απόψεις ε, των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Αλλά έχουμε διάσταση απόψεων ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλες αυτές οι διαφορές καταδεικνύουν κυρίως δύο τεινά. Το πρώτο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συνένεση είναι δυνατή μόνο ως προς την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να βρούμε συνένεση όπως ε, φάνηκε κατάφορα ε, επί τη συζήτηση της οδηγίας για την μητρότητα, είναι δύσκολο να βρούμε συνένεση για τον προσδιορισμό κοινωνικών πολιτικών που διασφαλίζουν κοινωνικά δικαιώματα. Μακάρι να κάνουμε λάθος, μακάρι να γελιόμαστε και μακάρι να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο για να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε αυτά τα δικαιώματα και τη βελτίωση των συνθήκων για να εξισορροπηθεί ο επαγγελματικό με τον ιδιωτικό βίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φάνηκαν ήδη κατάφορα οι μεγάλε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών στην προσέγγιση του στα ζητήματα αυτά. Ήδη και σήμερα στη συζήτηση το καταλάβαμε. Οπότε θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε στη ένταξη σε οποιαδήποτε τελικά οδηγία ε, τη ρήτρα της μη υποβάθμισης των κατοχυρωμένων δηλαδή δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, για παράδειγμα, οι προτινόμενες προτάσεις, αν εφαρμοστούν στην Πορτογαλία και υπερισχύσουν της εθνικής νομοθεσίες, θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των ε, κατοχυρωμένων σήμερα κοινωνικών δικαιωμάτων στην Πορτογαλία. Επίσης, για τις περιόδους της και τι διάρκειε τη άδεια. Θεωρούμε ότι η διάρκεια τη άδεια θα πρέπει να έχουμε μια ανωδική τάση και για την ε, μητρότητα και για την πατρότητα και για την γονική άδεια. Να υπάρχει μια τάση ε, επιμήκυσης ε, της διάρκεια και επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του παιδιού, τη γυναίκα, αλλά και στο ζευγάρι και στο, στην μονάδα την οικογενειακή που προσδιορίζουν. Επίση, να λάβουμε υπόψη και τι στάσει διεθνών οργανισμών. Μην ξεχνάτε τη σύσταση τη Παγκόσμια Οργάνωση ε, Υγεία, που λέει ότι το πρώτο εξάμεινο ε, για τα παιδιά ε, συστήνεται αποκλειστικό θυλασμό. Και αυτές οι συστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να προσδιορίσουμε τις, διάρκειες, τις κατάλληλες διάρκειες των διαφόρων αδειών. Επίσης, αυτή η η περίοδος της άδειας, η διάρκεια της άδειας, κυρίως της γονικής άδειας, θα πρέπει ε, να απορρέει από μία ευθύνη του ζευγαριού και να υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να εξασφαλίσουμε ή να βελτιώσουμε τις άδειες ε, τις γονικές αν η αποδοχές της άδειας δεν ε, είναι ίσες με τον πλήρη μισθό το επίπεδο θα είναι, πρέπει να είναι 100%. Επίσης δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη γέννηση με μία αρρώστια. Και όλες αυτές οι εξομοιώσεις με την αρρωτική άδεια νομίζω ότι είναι γελίες. Επίσης, ε, οι απολαβές ε, σε περίπτωση γονικής άδειας θα πρέπει να είναι το 100% του μισθού. Η δεμή θα... Ε, είναι σαν να τιμωρούμε τον, το ζευγάρι ή τη γυναίκα ή όποιο βγαίνει στην άδεια. Και ούτω ή άλλω οι γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν κατά 17% λιγότερο από τους άνδρες. Οπότε αν δεν έχουμε πλήρη ε, αμοιβή στη διάρκεια, πλήρη αποζημίωση, πλήρης αποδοχή στη διάρκεια της, αγωνικής άδεια, θα μειωθεί αισθητά ο προπολογισμό ε, του ζευγαριού του νοικοκύριου είμαστε κατά οποιασδήποτε άλλη ε, λύση ε, με χαμηλότερο ποσοστό. Και με την πλήρη κάλυψη, το 100% θα δώσουμε κίνητρα και στου άνδρε για να διεκδικήσουν αυτό το άδεια τη άδεια πατρότητα. Και στην Πορτογαλία ισχύει, ακριβώ επειδή υπάρχει δυνατότητα μεταβίβαση, έχουμε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό άδεια πατρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά το ποσοστό για τι αποδοχέ είναι 100% του μισθού. Επίσης, αυτές ε, οι άδειε θα πρέπει να μέσως μετά τη γέννηση του παιδιού η γονική άδεια και όχι να επεκτείνεται 10-12 μήνες μετά τη γέννηση. Επίσης, υπάρχει μια της γονικής άδειας με την άδεια για την παροχή φροντίδα στην οικογένεια. Και μάλιστα αυτή η έννοια στην πορτογαλική νομοθεσία κατοχυρώνεται και υπάρχει δυνατότητα 30 μέρες το χρόνο άδειε για την παροχή φροντίδας σε κοντινούς συγγενείς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συγχαίουμε αυτέ τι έννοιε τη γονική άδεια με την άδεια για την παροχή φροντίδα σε κάποιο μέλο οικογένεια. Ό,τι αφορά την παροχή υποδομών στήριξη, δηλαδή βρεφονιπιακών σταθμών, κέντρων ε, φύλαξη και ε, φροντίδα, ε, αυτά προποθέτουν δημόσια κονδύλια και δίκτυα που θα εξυπηρετούν αυτές τις υποδομές ε, ε, παροχής φροντίδας και φυσικά να έχουμε δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στις υποδομές αυτές για να μην επιβαρυθούν επιπλέον ε, οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά κατακλείδη, έγινε λόγος για την ελαστικότητα στις ρυθμίσεις της εργασιακές η ενσωμάτωση της αρχής της ευελιξίας δεν θα πρέπει να ε, θεωρηθεί ως πρόσχημα για να διευκολύνουμε τάχα την ε, ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Αυτό που θα πρέπει να ε, προτάξουμε είναι κυρίως προσαρμογή της, του ωραρίου εργασίας στην, στις ανάγκες της οικογενειακές του πατέρα της μητέρας και θα πρέπει να μειωθεί το ωράριο εργασίας. Αυτό το περισσότερο να είναι το ζητούμενο και όχι ε, επιμερισμό στη διάρκεια της εβδομάδας ή κατανομή στη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν καταλαβαίνουμε αυτό που λένε μερικές επιχειρήσεις ότι η μητρότητα τους δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό είναι αδιανόητο. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ποσοστό ενεργείας υψηλό γύρω στο 8%, 18% ε, σε μερικές χώρες. Επίσης, Έχουμε συνθήκες ορισμέ, ε, ε, συμβόλαια εργασιακά ορισμένου χρόνου και όχι αορίστο αυτό είναι ο κανόνας. Δεν είναι πρόσφορες συνθήκε για τη λήψη άδεια και ούτως ή άλλως κάθε επιχείρηση έχει ένα εξάμεινο για να προετοιμάσει και να προλάβει ε, να προετοιμαστεί για την απουσία του γονιού γιατί δεν γίνεται μέσα μια νύχτα η εγκυμοσύνη, δεν εκπεραιώνεται. Οπότε έχει τουλάχιστον έξι μήνες η επιχείρηση να προετοιμαστεί και να λάβει τα μέτρα της ε, για να καλύψει αυτή την απουσία. Θα μπορούσε να δώσει ε, συμβόλαια περιορισμένα για το χρόνο αυτό κατά το οποίο θα απουσιάζουν οι γονείς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιους μηχανισμούς κοινωνικής και εργασιακής προστασίας φυσικά ε, για τις γυναίκες ε, είναι αυτονόητο, αλλά και για τους άνδρες, για να μπορέσουν να απολαύσουν και στην πράξη δικαιώματα που θεωρητικά κατοχυρώνονται στην νομοθεσία. Επίσης, δεν αρκεί η νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων, γιατί αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου για την εγγύηση και την πρακτική απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων, τότε θα μείνουν στα χαρτιά απλώ και δεν θα εφαρμόζονται στην πράξη. Στην Πορτογαλία δυστυχώς έχουμε όλο και περισσότερες ε, περιπτώσεις γυναικών και ανδρών που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν, να απολαύσουν τα δικαιώματα που είναι νομοθετικά ε, καταχειρωμένα γιατί φοβούνται ότι αν ε, τα αντεκδικήσουν θα χάσουν την δουλειά τους. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Στο πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον David Κάσα για την πολύ ισόρροπη προσέγγιση. Συμφωνώ και εγώ ότι χρειαζόμαστε αξιοπρεπή αμοιβή τη γονική άδεια. Το δείχνουν όλε οι μελέτε. Ο βασικό λόγο για τον οποίο δεν παίρνουν άδεια ε, οι πατέρε γονικοί είναι ότι δεν πληρώνονται σε κανονικό επίπεδο και σε αξιοπρεπές. Για να τους αθαρρύνουμε λοιπόν θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό, να το αναθεωρήσουμε. Ευέλικτες μορφές εργασίας. Δεν είναι εύκολο πάντα να ε, φέρει ισορροπία αυτό. Κάποιος συνάδελφος από τους σοσιαλιστές είπε ότι θα πρέπει να έχουν ευέλικτη διαχείριση του χρόνου ε, οι ε, εργαζόμενοι χωρίς να ε, να κινδυνεύει η επιβίωση της εταιρεία. Η επιβίωση νομίζω αυτό είναι υπερβολικό. Οι εταιρείε θα πρέπει να είναι και κερδοφόρες και ανταγωνιστικές. Οι μεγαλύτερες εταιρείε έχουν περισσότερες δυνατότητες. Σε, ήδη υπάρχει ευελιξία ε, στην εργασία ε, στις πολύ μεγάλες εταιρείες. Για τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζω να έχουμε λοιπόν εκεί και αναλογικότητα και ισορροπία. Ο Άνταμ Κόζα μίλησε για την ανάγκη να ε, ε, διατηρήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας την εθνική νομοθεσία και ο συνάδελφος από την Πορτογαλία είπε ότι δεν θα πρέπει τίποτα σε αυτή την οδηγία να χαμηλώνει κάποια στάνταρ και προδιαγραφές που έχουν τα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε πολύ από εμά τι έγινε με την οδηγία για την άδεια μητρότητας και το τελευταίο που θέλουμε είναι να το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στη συγκεκριμένη πρόταση. Με όλες αυτές λοιπόν τις επιφυλάξεις θα πρέπει να παρατηρούμε και να κοιτάξουμε και την ε, εθνική νομοθεσία για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ιρλανδία, που ακούσαμε τι έγινε στην Ιρλανδία, εμείς έχουμε ήδη άδεια για τους φροντιστές. Το 80% της φροντίδας στην Ευρώπη είναι άτυπη, είναι οικογενειακή φροντίδα, 75% ε, μάλιστα των φροντιστών είναι γυναίκες. Για ποιο λόγο ε, έχουμε την ευτυχία να ζούμε περισσότερο όλοι μας και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται κάποια φροντίδα ειδική. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία και στα πλαίσια αυτά πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία χρειάζεται ακριβώς για να βοηθήσει και να ε, υποστηρίζει. Άκουσα κάποιους συναδέλφους να λένε ότι δεν είναι σωστό το ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω αρμοδιοτήτων διαφωνώ έντονα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά στη συγκεκριμένη έκθεση. Πάντως είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η οικονομική υποστήριξη δεν είναι αρκετή πάντα. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε ε, μακροπρόθεσμη φροντίδα, φύλαξη των παιδιών, δομές μόνιμες, ουσιαστικές για να υπάρχει πραγματική ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και για τους γονείς και για τους φροντιστές. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και καταρχήν ε, έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Συμφωνώ για τα ωραία ηλικία, για παιδιά με ειδικέ ανάγκες, αναπηρίες, για έκτακτες περιστάσεις. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Και τέλος, το είπαν ε, ένας-δύο συνάδελφοι, το θέμα των συντάξεων. Πολλές φορές ε, όσοι φεύγουν από την εργασία τους και απουσιάζουν για ε, να φροντίσουν κάποιους, ε, χάνουν μισθό, χάνουν εισοδήματα και δεν καταβάλουν εισφορές και τελικά είναι χαμηλότερε οι συντάξει μετά από 30 χρόνια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι σημερινοί φροντιστές δεν θα γίνουν οι αυριανοί ε, φτωχοί ηλικιωμένοι και κυρίως φτωχές ηλικιωμένε γιατί πρόκειται για γυναίκες ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, χαίρομαι για την προσπάθεια αυτή, συγχαρητήρια στον εισηγητή και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ κυρία Σόιτροβα. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εξαγητή, οι προτάσεις του είναι πολύ λογικές, ισορροπημένες. Και μας απασχολεί να προστατεύσουμε το συμφέρον των γονιών, των παιδιών, των φροντιστών. Η παροχή καλής ποιότητας ε, υπηρεσίας προσφερόμενης στο παιδί ως προσέγγιση μας φαίνεται καλή, η προσήκουσα, το προσήκον εισόδημα. Για να είναι προσήκον δεν μπορεί να έχει αναφορά στο επίδομα ή στην ε, ε, αποζημίωση για άδεια ασθενείας. Για τις μητέρες τουλάχιστον. Ε, για τους πατέρες θα μπορούσε γιατί υπάρχει αντιστοιχεία αυτή με τη μητρική άδεια. Ωστόσο πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό για την άδεια ε, επί του ακαθάριστου εισοδήματος. Για το ελάχιστο ποσοστό επίσης έχω κάποιες παρατηρήσεις. Ένα 75% θα πρέπει να είναι μάλλον υψηλό. Ως κατώτατο επίπεδο μας λέτε 75% θεωρώ ότι είναι υψηλό, θα πρέπει να έχουμε κάποια εναλλακτική. Ο εισηγητής στοχεύει στην προστασία των μικρομεσαίων, συμφωνούμε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βεβαίως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι ευέλικτα στο προσδιορισμό του γραφειοκρατικού βάρους, της γραφειοκρατικής επιφάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενότατη ηλικία. Ο εισηγητής προτείνει 10, η Επιτροπή 12. μπορούμε να είμαστε πιο γενναιο... μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά, διότι νομίζω ότι τα 8 χρόνια φτάνουν ναι. για να καλυφθεί ο στόχος της οδηγίας. Κάποια άλλα θέματα πρέπει να καλυφθούν. Καταθέτω τροπολογίες για την άδεια φροντιστή που είναι σχετικά ε, στενός ορισμός της θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τουλάχιστον τα κράτη-μέλη να ανοίξουν το πεδίο ώστε να μπορεί κανείς να φροντίσει περισσότερους συγγενείς. Η μη μεταφερσιμότητα καλή, αλλά για τους τέσσερις μήνες νομίζω ότι είναι υπερβολικός ο περιορισμός στο να μην υπάρχει μεταφερσιμότητα. Όπως είπαν και κάποιοι συναρφοί για τις μικρομεσαίες, πάλι θα είναι δύσκολο περισσότερη ευελιξία για τον γονεί. Ε, μια πιο σύντομη περίοδο λοιπόν με μεταφερσιμότητα θα πρότεινα εγώ και εναλλακτικά θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να προσφέρουν συμπληρωματική γονική άδεια για όσους γονείς μοιράζονται τα οικογενειακά βάρη και τη φροντίδα των παιδιών που θα ήταν και ένα καλό κίνητρο. Ξέρω ότι αυτό, ειδικά στη Γερμανία, φέρνει αποτελέσματα. Θα καταθέσω τροπολογίες και είμαι βεβαίω ότι θα έχουμε μια καλή έκθεση για ε, συμφωνία τελικά στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Κύριε Κάσα, εσείς, όχι, να ρωτήσω την Επιτροπή, αν είναι κάποιος εδώ που θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Ολιβιέ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μου και την μεγάλη εκτίμηση μου και αναγνώριση του έργου. Κυρίως για την άδεια πατρότητας με πλήρη αμοιβή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή στην αγορά εργασία και πιστεύω ότι οι προτάσει αυτέ συμβάλλουν προ αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι φορά την επικουρικότητα, υπάρχει ήδη πρωτοβουλία ευρωπαϊκή για, την, για το συνδυασμό ε, επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στις διάφορες πολιτικές. Κάτι που δείχνει την ανάγκη ευρωπαϊκής δράσης εδώ, που ευθυγραμμίζεται και με την αρχή της επικουρικότητας. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ελάχιστο κοινό επίπεδο, τουλάχιστον για την αγωνική και άδεια πατρότητας, θα βελτιώσει τη διαφάνεια της πρότασης και της αφήνειά της. Και τέλος, δεν συμφωνώ με την προτινόμενη μνήμα της εθνικής νομοθεσίας. Αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς σε συλλογικές συμφωνίες και πάραξ πρακτικές για τον ορισμό του εργαζομένου. Σίγουρα κάτι τέτοια μνήμα αφήνει την, να εννοηθεί ότι υπάρχει διακριτική ευχαίρεια για τον ορισμό του εργαζομένου στα κράτη-μέλη, κάτι που είναι παραπλανητικό και επιτείνει την έλλειψη ασφάλειας δικαίου, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Ευχαριστώ και τώρα λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κάσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερο που οι σκιώδεις ηγητές μας και οι λοιποί συνάδελφοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης γενικώ και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στην πρόταση, πρόταση αυτή και ταυτόχρονα να είμαστε και ρεαλιστές. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά για την πρόταση αυτή. Σημείωσα όλες τις προτάσεις και κυρίως την ε, ιδιαίτερη μερίμνα για τους γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες. Θα δούμε πώς θα μεριμνήσουμε ιδιαίτερα για αυτούς. Για την ε, Βρετανική νομοθεσία θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, και για την Πορτογαλική νομοθεσία να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε τη ρήτρα της μη υποβάθμισης στην πρόταση, ώστε οι χώρες που έχουν πιο ευνοϊκούς όρους για τις περιπτώσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν ε, οφείλουν να τους υποβαθμίσουν λόγω της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης. Επίσης, μην ξεχνάτε την ιστορία που είχαμε με την άδεια μητρότητας. Γιατί αν δείξουμε ρεαλισμό θα έχουμε μία από τα ίδια και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί ε, η ιστορία που έγινε με την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στο ρεαλισμό σας και να βοηθήσουμε ε, την άδεια μητρότητας να την ε, εγκρίνουμε και να ξεκινήσουμε με κάτι ρεαλιστικό με τη συγκεκριμένη πρόταση γιατί δεν θα είναι εύκολο οι διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο. Γι' αυτό εμείς είμαστε, ας μην είμαστε υπερβολικοί εμείς σε ό,τι αφορά την υποβολή νέων προτάσεων και τον υπερβολικό εμπλουτισμό της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την τροποποιήσουμε μεν, αλλά με ισορροπημένο τρόπο. Δεν πρόκειται εμείς να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου ή όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο ας συμφωνήσουμε σε ελάχιστες κοινέ προδιαγραφές. Θα είναι μία αρχή που θα μας βοηθήσει όμως να βελτιώσουμε στο μέλλον την νομοθεσία μας και κυρίως την οδηγία για την άδεια αργότερα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ όλους σας για τη συζήτηση αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 13 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Εδώ θα το εγκρίνουμε στις 11 Ιουλίου και στην Ολομέλη αποθέτω μετά τις 9 διακοπές. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό ακόμα. Μην το δέσετε κιόλα. Άρα, φτάσαμε εσύ στο τελευταίο θέμα για σήμερα στη Μέση Διαταξή. Καταστατικό επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι του κυρίου Μπέκερ. Και με έχει εντυπωσιάσει το γεγονό ότι έχουν παραμείνει τόσοι πολλοί συνάδελφοι παρόντε σε αυτή την προκεχωρημένη ώρα για να σα ακούσουν. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Μπέκερ, ευχαριστώ και του συναδέλφου που έχουν λίγο χρόνο ακόμα να μα αφιερώσουν. Και ευχαριστώ για όλου του κοιόδη ηγητέ για την αγαστή συνεργασία και τον κύριο Μαστάλκα που είναι αρμόδιος επί της ουσίας στην Επιτροπή Γιούρι. Ε, και το EPRS ε, για την εξαιρετική μελέτη ε, που μας υπέβαλε. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικές στην ευρωπαϊκή οικονομία με αμύωτη ανάπτυξη. Από το 2008 και μετά ακόμα και επί της κρίσης υπάρχει ανάπτυξη παρέχουν υπηρεσίες ε, απασχολώντας 10% του συνόλου των εργαζομένων αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Και από την αρχή της κρίσης και μετά έκαναν και προσλήψεις 1,8 εκατομμύρια εργαζομένων. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα βοηθάει την κοινωνική ένταξη ε, ε, μειονεκτούν των ατόμων, δίνουν κοινωνικές υπηρεσίες, προστατεύουν το περιβάλλον. Αυτά τα δύο δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Γι' αυτό και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι απαραίτητο έτσι ώστε η οικονομία της αγοράς να γίνει έτη κοινωνικότερη, γιατί είναι τμήμα της οικονομίας αγοράς και οι κοινωνικές επιχειρήσεις και εταιρείε. Γι' αυτό θέλουμε ένα καταστατικό επιχειρήσεων κοινωνικής ε, οικονομίας είναι ενώσεις, είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως ο Ερθρός ε, Σταυρός, ε, ιδρύματα και συνεταιρισμοί. Όλο και περισσότερο γίνεται σημαντική αυτή η μορφή επιχείρησης γιατί είναι ελκυστική για τους νέους ε, που έχουν ιδανικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θέλουν να τα κάνουν πραγματικότητα. Τα κεντρικά σημεία λοιπόν της δικής μου γνωμοδότησης ποια είναι. Πρώτον, ναι στα κέρδη, αλλά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ε, υπάρχει προϋπόθεση σε ε, μεγάλο βαθμό και κατά μεγαλύτερο κλάσμα να επανεπενδύονται τα, τα κέρδη αυτά για να εξυπηρετούνται ακόμα περισσότερο και καλύτερα κοινωνικοί στόχοι. Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ε, φέρνουν την απόδειξη ότι έχουν πραγματικά κοινωνική δράση και επίδραση στο εσωτερικό της αγοράς. Επίσης, είναι πάρα πολύ καλό να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές τη κοινωνικής οικονομίας είναι επιχειρήσεις που έχουν ορατά αποτελέσματα. Αν δούμε τι είδους εταιρείε είναι αυτές, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει ξενοδοχείο της Κάριτας και μάλιστα ε, μια ε, υπηρεσία, ένας οργανισμός που διοργανώνει εκδηλώσεις. Και πού είναι το κοινωνικό. Το κοινωνικό είναι ότι η Κάριτας απασχολεί και εργοδοτεί ε, μακροχρόνιους ανέργους. Δηλαδή είναι υψηλή αξίας κοινωνική προσφορά. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι βγαίνουν από την κατάσταση την δινή στην οποία έχουν πέρα. Ή υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις ε, που επιδιορθώνουν ε, τηλεοράσεις ή ποδήλατα και ποια είναι η κοινωνική προσφορά. Δεν υπάρχει κοινωνική προσφορά, αλλά οι εργαζόμενοι είναι προεγκρατούμενοι ε, που έχουν ε, αποφυλακιστεί. Και πάλι λοιπόν ε, είναι τεράστιος ο κοινωνικός αντίκτυπος. Για να μην πω ότι κάνουν και οικονομίες από τους προπολογισμού για τα κοινωνικά επιδόματα των κρατών μελών μας. Πόσο μάλλον που αποκτούν ένα κοινωνικό ρόλο οι άνθρωποι αυτοί και μια σημασία, ένα νόημα στη ζωή τους όταν μπορούν να έχουν ε, τέτοιε δραστηριότητε. Α πούμε, υπάρχουν κάποια διαγνωστικά κέντρα για τον καρκίνο του μαστού, όπου οι ψηλαφίσει για την εξέταση αυτή γίνονται από τυφλού, παρακαλώ. Και δεν χρειάζεται να σας πω ότι όλες εκείνες οι επιχειρήσεις ανήκουν εδώ ε, ε, ε, που δραστηριοποιούνται στη φροντίδα, στην υγεία, στην περίθαλψη, στην φύλαξη των παιδιών. Και αυτοί οι κοινωνικοί σκοποί εξυπηρετούνται από αυτές τις επιχειρήσεις και δεν χωρά καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Στην έκθεση μας λοιπόν στην γνωμοδότηση ζητούμε ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μια πρόταση που δεν είναι ακόμα συνενετική, δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά να σας την αναφέρω. Να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης όπου οι κοινωνικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν ένα σήμα, ένα πιστοποιητικό της κοινωνικής επιχείρησης. Για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό. Για να προσελκύονται ιδιώτες επενδυτές σε αυτή την κοινωνική οικονομία. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι αυτές στην Ευρώπη. Και ένας επενδυτής δεν μπορεί να ελέγξει εάν ε, πραγματικά είναι κοινωνική επιχείρηση και αξίζει το όνομά της. Αν, αν θέλουμε λοιπόν χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα, θα τα βρούμε από εκείνους τους επενδυτές που δεν θέλουν τη μεγάλη απόδοση των χρημάτων, αλλά θέλουν να έχει ένα κοινωνικό σκοπό που να επιτελεί. Για να γίνει αυτό να το εξασφαλίσουμε χρειάζεται ένα σύστημα πιστοποίησης. Και τελευταίο, χωρίς αυτό βέβαια να είναι το λιγότερο σημαντικό και πάρα πολύ σύντομα, παρακαλώ μέχρι σε 9 Απριλίου, 5 ώρα το απόγευμα, να κάνετε τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Becker. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Κύριος Παύλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη του κυρίου Λόπε, του συναδέλφου που δεν μπορεί να έρθει εδώ, διότι έχει μια ε, δέσμευση με τα Ευρωπαϊκά Σωματεία στη Γανδία. Η θέση του λοιπόν ως και όδος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Καταρχάς ευχαριστούμε όλους για τη δουλειά που έκαναν και τον εισηγητή μας και από τη Γιούρη και από την Έμπλη νομοθετική πρωτοβουλία και συντονισμός μεταξύ συναρμόδιων επιτροπών. Ο εισηγητής μας πολύ σωστά εξετάζει τις συστάσεις από την ε, μελέτη ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας του υπερές που ανέφερε και ο εισηγητής, η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρχει ε, σχεδιασμός και σύσταση ενός συστήματος ε, με προδιαγραφές για κάθε εταιρεία που μπορεί, η επιχείρηση που μπορεί να προσφέρει κοινωνικό έργο εξαρτήτως της νομικής φύσης της. Και έτσι πρέπει να είναι ένα σύστημα, μας λέει ο εισηγητής, το οποίο θα μπορεί θελοντικά να συμμετέχει μια επιχείρηση με κριτήρια και προϋποθέσεις ε, για την διατήρηση του χαρακτηρισμού ως ε, επιχείρησης κοινωνικής ε, υπηρεσίας και ελληνικής οικονομίας και αλληλεγγύης. Η χρηματοδότηση, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει πολύ μεγάλη σημασία και συμφωνούμε γενικά με τις προτάσεις του εισηγητή, της ΕΜΠΛΗ. Θεωρώ τις πάντως ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροπολογίες που θα έχουν την εξή κατεύθυνση. Θα πρέπει να ενισχυθεί η έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνήσει ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ξεπερνά την απλή επισήμανση ή ε, πιστοποίηση. Θα βοηθήσει και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Στρατηγικές στόχοι θα πρέπει να είναι τα κριτήρια. Πρέπει να έχουν πραγματικά όρους υπηρεσίας κοινωνικής αυτές οι επιχειρήσεις και αυτό να αξιολογείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και ίσως θα ήταν καλό να επισημανθούν και κάποια μέτρα για την πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων σε δημόσιες προμήθειες και δημόσιες αγορές. Πρέπει να βρούμε τρόπους να προαγάγουμε το αξιόλογο έργο αυτών των επιχειρήσεων μέσα από τον ορίζοντα 2020, γιατί και καταπολεμούν την ανεργία και προάγουν την ανάπτυξη και βοηθούν στην εξάλληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι καλή δουλειά που έχει κάνει ο τον ευχαριστούμε. Είμαστε στα θέση του για συνεργασία με τις πολιτικές προτάσεις που θα καταθέσουμε με βάση βέβαια τις ανάγκες του τομέα αυτού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάκιντάιρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και επιτρέψτε μου καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη Γιάννα που είναι σκιώδη συγγεντρία και δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Θα ήθελα πάντως να ευχαριστήσει τον εισηγητή, όχι μόνο για την πρόταση, αλλά και για τη διάθεση να ε, αφουγκραστεί τους άλλους σκιώδη οδησηγητές και να συζητήσει μαζί τους. Οπωσδήποτε είναι αξιόλογη πρωτοβουλία της υποστήριξης των επιχειρήσεων με, της κοινωνικής οικονομίας και αυτός είναι και ένας τρόπος να δώσουμε απάντηση στις ανάγκες των ε, τοπικών ομάδων πληθυσμού και κοινωνίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές φορές έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς έντασης εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στόχος της Γιάννας είναι να υπάρχουν κριτήρια σωστά, όπως είπε και ο εισηγητής ε, πολύ σωστά, οι τυπικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι στο δυνατόν λιγότερες για την εξασφάλιση της πιστοποίησης και για να θέλει καλύτερη συμμετοχή και των ε, κοινωνικών αυτών επιχειρήσεων σε δημόσιες συμβάσεις, χωρίς βέβαια να υπάρχουν και στοιχεία θέμη του ανταγωνισμού σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις. Ωστόσο, θέλει να υπογραμμίσει για να ότι μερικές φορές παραγνωρίζεται η σημασία της ε, ε, εξασφάλιση από αυτές τις επιχειρήσεις ενός ε, υγιούς επιχειρησιακού περιβάλλον. Βέβαια ξέρω ότι αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν γνωρίζεται η σημασία αυτή το, με τον ίδιο τρόπο και θα το σεβαστεί. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για καλά αποτελέσματα. Και αν μου επιτρέπετε τώρα να περάσω σε μια προσωπική παρατήρηση, σε κάποιε προσωπικέ παρατηρήσει. Με μεγάλη χαρά ξαναβλέπω το Χάιντ Σπέκια στο θέμα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Είναι ε, μεγάλος αγωνιστής των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των ε, επιχειρήσεων κοινωνική οικονομίας και θέλω να πω ότι και εγώ που είμαι πολύ περήφανη που είμαι διευθύντρια Λεμένα Βασίλειο σε με μια, σε μια επιχείρηση που ε, στην παραγωγική της διαδικασία χρησιμοποιεί κοινωνικά ε, ε, επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο αυτό και μπορούμε να το κάνουμε όλοι έτσι ώστε να προσφέρουμε ε, κέρδος και στην κοινωνία γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα της πιστοποίησης ώστε και ο πολίτης να γνωρίζει ότι όταν αγοράζει αυτά τα προϊόντα και υποστηρίζει την συγκεκριμένη μάρκα της, του εμπορικό σώμα της επιχείρησης θα υποφελούνται και οι συμπολίτε του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χάρκη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την πολύ αξιόλογη προσπάθειά του και να συμφωνήσω και μαζί του και με τους προλαλήσαντες στο, ως προς τον πολύ θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τέτοιες ε, επιχειρήσεις ε, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Πολύ σωστά ζήτησε το κοινωνικό σήμα ως μέθοδο και όχι το ευρωπαϊκό νόμιμο ε, πρότυπο, λογότυπο μάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μιλήσει για τέτοια ε, εταιρεία για το 2006 και το 2012 πρότεινε ένα καταστατικό για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Αλλά και οι δύο προτάσεις αποσύρθηκαν στη συνέχεια, γιατί δεν ε, είχαν συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη. Ευχαριστώ λοιπόν τον Ρίση, γιατί υποκολούσε διαφορετική πορεία και όχι την νομικά δεσμευτική ε, νομική μορφή. Ε, σε ό,τι αφορά το δικό μας ψήφισμα το 2015 για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, εκεί απευθύναμε έκκληση ε, στην διευκόλυνση της πρόσβασης στις κρατικές προμήθειες και την βελτίωση στην δανειοδοσία. Ε, δεν θυμάμαι αν μπήκε τελικά το κοινωνικό σήμα στο τελικό κείμενο, πάντως σίγουρα το είχαμε συζητήσει. Εγώ είμαι υπέρ ενός κοινωνικού σήματος και συμφωνώ ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αξίζει το σήμα, τουλάχιστον το χαρτί πάνω στο οποίο είναι γραμμένο. Και επίση να διευκολύνουμε την πρόσβαση στι δημόσιε συμβάσει. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Και η Άθεα ναι, είπε για τη θέση τη και οδησηγήτρια κυρία Ζετινάσκα, που λέει θα πρέπει να φροντίσουμε και για τι υπόλοιπε επιχειρήσει, να μην υπάρχει ε, αθέμητο ανταγωνισμό ει βάρο του. Πάντω, έχουμε ήδη στην νομοθεσία μα για τι ε, δημόσιε συμβάσει και τι κρατικέ προμηθείε διάφορα επίπεδα και βαθμού πρόσβαση. Οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα εδώ. Και επίση συμφωνώ με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση. Και θα έλεγα και προσβλέπω σε πραγματικά μεγάλο αριθμό τροπολογιών στην ε, έκθεση αυτή. Κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά, κύριε Μπέκερ, γιατί πιστεύω ότι η έκθεση θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη και να βελτιώσει το κοινωτικό πλαίσιο. Γιατί είναι απαραίτητο να θαρρύνουμε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Συμφωνώ με την πιστοποίηση, γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη. Επίσης, θα πρέπει η πρότασή μας να επιτρέπει στα κράτη-μέλη μια μεγαλύτερη ευελιξία στις δράσεις τους. Ελπίζω το πλαίσιο που θα διαμορφώσουμε να στηρίξει κάποιες πρωτοβουλίες των κρατών μελών σχετικά. Και είμαι υπέρ, επαναλαμβάνω, της έκθεσης. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κλάινς από τη Γενική Διεύθυνση Growth της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρόν ακόμη. Αν θέλετε το λόγο, πολύ ευχαριστώ κύριε Κλάινς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμότατα για τη συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως σημαντική προτεραιότητά την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ε, και εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαστε με την ε, ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών νομικής και οικονομικής υποστήριξης για να στηρίξουμε την ε, προώθηση της κοινωνικής και ελληνικής οικονομίας στην Ευρώπη. Είχαμε και την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που συνεχίζει τις εργασίες της. Το 2013 διεκπαιρεώσαμε μία μελέτη με θέμα τη χαρτογράφηση του είδους των δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας μας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Και κατά τη χαρτογράφηση αυτή, ε, στόχος μας είναι να αναδείξουμε κάποια εθνικά συστήματα επισήμασης ε, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν. Έχει ε, γίνει και μια επικαιροποίηση της έκθεσης, οπότε η ενημερωμένη έκθεση θα σας θετεθεί στα τέλη ε, του τρέχοντος και σε αρχές του επόμενου έτους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω των, ε, του ΕΦΣΥ, του Κοινωνικού Ταμείου, των Διαρθρωτικών Ταμείου και της πρόσβασης κρατικών και ιδιωτικών επενδυτών ε, σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης σημαντικό είναι ότι οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι υπέρ και ασχολούνται με την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος με συμβασμό όμως των διαφόρων προσεγγίσεων και παραδόσεων των κρατών μελών. Ε, έτσι έχει φανεί από κάποια θετικά παραδείγματα. Ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σήμα θα πρέπει να εμπλέξει ενεργά όλους τους ε, ενδιαφερόμενους και σε τοπικό και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Γιατί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι αυτοί που είναι πλέον ευαισθητοποιημένοι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά έχουν και την δυνατότητα να είναι οι υπέρμαχοι και οι προτεργάτες της αλλαγή στην οτροπία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ο συγητής, παρακαλώ, αν θέλετε να πείτε τίποτα. Äh, Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι εκ των προτέρων για την προθυμία σας να καταθέσετε τροπολογίες για να εμπλουτίσετε και να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την παρούσα γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ για τα ειλικρινή λόγια και τα ενθαρρυντικά ε, των κυρίων Μακεντάερ, Χάρκιν και άλλων συναδέλφων. Και με μεγάλη χαρά έξω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας επιβεβαιώνω, ως ε, εισηγητής ε, της, ε, κοινωνικής, ε, της πρωτοβουλίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, επί Επιτρόπου Μπαρνιέ ακόμα, ε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προεργασία που έχει γίνει και χαίρομαι που θα τα αξιολογήσετε και πάλι για να βάλουμε άλλο ένα λιθαράκι εδώ για να ενισχύσουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ε, ευχαριστώ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 9 Απριλίου στις 5 ώρα το απόγευμα. Η έγκριση εδώ θα είναι στις 17 Μαΐου, ενώ στη Γιούρη που είναι αρμόδια επί της ουσίας νομικών θεμάτων στις 20 Ιουνίου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ Σα σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Uh, Τουλάχιστον ε, όσοι παραμείνατε μέχρι τέλους. Λήξη συνεδρίασης. Yeah. It was an interesting debate uh, to the very end.